Ε, των οργάνων του. Καλωσορίσατε θερμά αγαπητοί συνάδελφοι. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα στη διάταξη των εργασιών. Θα ήθελα να σας πω ότι μετά τις συζητήσεις με τις πολιτικές ομάδες ε, θέλω να σας προτείνω αλλαγές στην ημερήσια διάταξη. Καταρχά, δήλωση του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας να προσθεθεί ως πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη σήμερα. Οπότε και οι ψηφοφορίες μετατίθενται για τις 7 αντί τις 6.30. Θα αρχίσουν στις 7 η ώρα οι ψηφοφορίες. Διαφωνεί κανείς? Όχι. Ούτω λοιπόν και εγκρίθηκε. Ευχαριστώ πολύ. Η διάσκεψη των Προέδρων, κυρίε και κύριοι, σήμερα ενέκρινε πρόταση για απόφαση ε, για σύσταση της ε, Ειδική Επιτροπής ε, με όνομα ΤΑΚΣ 2 που αντιστοιχεί με την προηγούμενη Επιτροπή ΤΑΚΣ 1. η απόφαση θα σας διαβιβαστεί και θα συμπεριληφθεί στις ψηφοφορίες προς ψήφιση. Ομόφωνα αποφάσισε έτσι η διάσκεψη των Προέδρων. Συμφωνείτε, διαφωνείτε. Ωραία, θα ψηφίσουμε συνέχεια για αυτή την Επιτροπή. Με αυτές τις αλλαγές, αν δεν ζητηθεί τίποτα άλλο, εγκρίνεται έτσι η μερίσια διάταξη. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Και ερχόμαστε λοιπόν στη συζήτηση για τη Σύνοδο κορυφη Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία.